Σαϊτής. Όντως και αυτή είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Η συζήτηση έληξε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία, εκθέσεις της κυρίας ε, Μπαραντίκα, του κυρίου Γκάλαχερ του κυρίου Γκρόμπερτσικ, του κυρίου Φερέιρα. Πρώτα μιλάνε οι συγκητές μας. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντζίκα για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρώτοι μου λόγοι θα είναι οι ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους του κλάδου της περιοχής. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα τόσο ώστε να πετύχουμε του στόχου μα. Θα πρέπει να υπάρχει επικεντρή δραστηριότητα και να μην τίθεται εν κινδύνο ο κλάδο τη αλληλεία. Και γι' αυτό θα πρέπει η βιομάζα του γάβρου να παραμείνει σε τέτοιο επίπεδο, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε τις, ε, κοινωνική και οικονομική κατάσταση που θέλουμε να πετύχουμε. Και έχουμε βέβαια κάποιε εκθέσει επιστημονικέ, και ούτω ώστε το ΤΑΚ περνάει και από τι πολιτικέ διαπραγματεύσει. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνεται η εκμετάλλευση και η αλλήλευση, ούτω ώστε τα, οι ποσοστώσει πρέπει να βασίζονται στι ε, επιστημονικέ εκτιμήσει για την βιομάζα. Τον Ιούλιο του 2009 κατεβάσατε κάποιε προτάσει. Αρχίσαμε τη δουλειά τον Σεπτέμβριο και είπαμε ότι θα πρέπει με του Γάλλου και τους ε, Ισπανούς και τους, τους, τους φορείς τους ε, να τα συμφωνήσουμε και να τα βρούμε σε σχέση με αυτά τα τα ύδατα και το Κοινοβούλιο στήριξε τι προσπαθειές σα υπήρξε συνένεση, λάβουμε υπόψη το ότι άρχισε να ισχύει συνήθεια της Λισαβόνας, υπήρχε αναφασιστικότητα ω προ το τι θα ισχύσει δυνάμει τη συνθήκης, Οπότε τον Νοέμβριο έγινε μια προστατοριστική ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας. Είχαμε ανοιχτή δουλειά όλοι συμμετέσχον και είχαμε διαφορετικέ αντιδράσεις από Συμβούλιο και Επιτροπή ετοιμάσαμε έναν ελεγκτικό κανονισμό ε, όμως δεν είχαμε αρκετές ε, πληροφορίες το οποίο μας οδήγησε σε κάποια ανασφάλεια, βεβαιότητα και πήραμε πρωτοβουλία ε, και η Ισπανική Προεδρία έγινε τριγωνικός διάλογος και απροσδόκητα μας είπε η Προεδρία ότι η αιτήση της Γαλλίας θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί το θέμα γιατί δεν είχαν συμφωνήσει για την νομική βάση. Μετά από τόση δουλειά παρέλυσαν όλα. Οπότε ρωτήσαμε τη νέα Προεδρία τι θα γίνει και απήντησαν ότι δεν θα πρέπει να βιάζομαι και να είμαι ανυπόμονη. Ε, επομένως, μια που δεν είχε βούληση. Λέτε πάρα πολύ γρήγορα ε, για τους διερμηνείς, κυρία Μπιλμπάου, λέει ο Πρόεδρος. Αν θέλετε, συνεχίστε. Αλλά όμως δεν γίνεται αντιληπτό αυτό το οποίο λέτε ολοκληρώθηκε χωρί να υπάρχει καμία συμφωνία, συνένεση, τριγωνικό διάλογο σε Ισπανική Προεδρία. Και οπότε ρωτώ την επομένη Προεδρία εάν επιθυμεί να συνεχίσει διαπραγματεύσει και μου είπαν ότι δεν θα πρέπει να βιάζομαι και να είμαι ανυπόμονη. Επομένω, ε, τώρα μια που θέλει το Συμβούλιο κάτι τέτοιο, προχωρήσαμε σε τέτοια ψηφοφορία, πήγαμε και στην νομική υπηρεσία, απορρίφθηκαν τρει τροπολογίε τη προσανατολιστική ψηφοφορία που ήταν πάρα πολύ βασικέ για τον κλάδο. Πρώτα-πρώτα, αυτό έχει σχέση με την ποσόστοση εκμετάλλευση και το 0,4 θεωρήθηκε καλό κατόπιν όσον αφορά τα ζωντανά δολώματα και τα τάκ είπαμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να μετράει ως αλίευμα και για τα, για τα τάκ και το άλλο θα, αυτό αφορά το, το, το αλίευμα γιατί θα πρέπει τώρα να δούμε πως η αξιόλογηση για τη βιομάζα θα ληφθεί υπόψη ή τότε πλήσονται διπλά οι, οι αλίες και με τα τάκ και με αυτή την αξιολόγηση. Εμεί θεωρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τη μείωση του 10% αλλά ποτέ κάτω από 7.000 τόνου. Οπότε, όσον αφορά το Κοινοβούλιο και τι αρμοδιότητέ του, αυτά το οποίο ισχύει είναι ότι οι Κομισιόν και οι Συμβούλιο δεν μα σέβονται. Και συζητούμε αυτή την πρωτοβουλία και μα ήρθαν νέα ανεπίσημα ότι ζήτησε το Συμβούλιο να αποσυρθεί η πρωτοβουλία. Αυτό ισχύει κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε να μας πείτε και να μα πείτε γιατί θα κάνετε. Θέλω σήμερα να μου δώσετε μια απάντηση. Επίση, θέλω η Βελγική Πρόεδρε να μου απαντήσει γιατί εζήτησε την απόσυρση της πρωτοβουλίας. Θέλω ξεκάθαρες σαφείς απαντήσει. 14 μήνε δουλεύουμε και καταλήξαμε μόνο σε μια ματέωση και σύγχυση και επομένω θα πρέπει να αποκτήσει η αξιοπιστική Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ο κλάδο έχει κουραστεί με τέτοιε μεθόδου και θέλει μόνο λύσει. Χάνουμε αξιοπιστία. Τουλάχιστον ε, αν, όχι να αυξήσετε την αξιοπιστία, ανακτήστε αυτή που χάσατε ε, από τότε που άρχισε αυτή η υπόθεση μέχρι τώρα. Ε, υπάρχει στην απόφαση και το, αυτό το, το προβλέπει η ψηφιακή τη Λισαβόνα. Ε, θα πρέπει να μας ε, σεβαστείτε και μόνο έτσι θα έχουμε τη ηγετικό ρόλο 21ο αιώνα και έτσι θα έχουμε και την διαφάνεια που θέλουμε. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε και εσείς αυτό το οποίο χρησιμοποιήσαμε και εμείς αυτές τις αρχές. Αυτό πάνω από την Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Ευχαριστώ κύριε Ο Κύριος Γκάλαχερ για τέσσερα λεπτά. I underline four minutes please. Uh, commissioner... Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου να ετοιμάσω αυτή τη σημαντική έκθεση ε, σχετικά με ε, το Σαφρίδι ε, και τα αποθέματα του και να ευχαριστήσω επίσης και τους εμπειρογνώμονες για την στήριξή τους. Χάρη στην στενή συνεργασία το διάλογο οι ιδέες των συναδέλφων μου επέτρεψαν να παρουσιάσω σήμερα αυτή την έκθεση και ελπίζω ότι θα γίνει δεκτός αποδεκτό. Η πρόταση αυτή βαθίζεται στο πρόγραμμα το οποίο συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εις την ε, διάσκεψη του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη το 2002 οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τα αλευτικά αποθέμωνα και στη συνέχεια ε, υπήρξε ένας κανονισμός ο οποίος ε, διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και οι μελέτες για το Σαφρίδι από το 1997 γίνονται ανατριετρία και αξιολογείται η κατάσταση των αποθεμάτων και στη συνέχεια διατυπώθηκε ένας τύπος για σχέση πλοίων με αλλιεύματα σαφριδιού που προβλέπει ένα τρόπο για να, φτάνουμε σε ένα ανώτατο επίπεδο σαφριδιού το οποίο ε, μπορεί να αλλιευτεί σε μια δεδομένη περιοχή και τα αποτελέσματα τα περιμέναμε για το 2009 αλλά έχουν καθυστερήσει. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να καθορίζει τις αλλιευτικές δυνατότητες ε, αλλά ε, μας πρότειναν μία πρόταση ε, η οποία όμως πρέπει να επιτρέπει ευελιξία και ε, να ε, καθορίζει το επιτρεπτό ε, ποσοστό και απορρίψεων αλλά και αλλιευμάτων και όχι να προφυλάσσεται απλώς το δικαίωμα του Συμβουλίου σύμφωνα με τις συνθήκες να καθορίζει τις δυνατότητες αλλιείας. Ε, θα ήθελα να πω ότι στην περιοχή του Βισκαϊκού υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε τις τροπολογίες του ΕΛΚ και της Ηνωμένη Αριστεράς διότι είναι ένα απόθεμα το οποίο καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Αν δεχθούμε την πρόταση του ΕΛΚ και της Ηνωμένης Αριστεράς, τότε το πρόγραμμα ε, θα αποδυναμωθεί γιατί θα χρειάζονται δύο προγράμματα για ένα απόθεμα. Οπότε θα ήθελα να σας ε, προτείνω να μην καταρτήσουμε ένα τέτοιο επικίνδυνο προηγούμενο για ένα πρόγραμμα διαχειρίσεως της αλληλείας σαφριδιών. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν κάτι τέτοιο θα το πράξουν μόνο για προσωπικούς λόγους και για λόγους που ε, ε, καλύπτουν τα κράτη-μέλη τους. Αλλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε ευρύτερα. Έχουμε Ισπανούς και Πορτογάλους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ανησυχίες και αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες τους και τις αντιμετωπίζω ή στο άρθρο 7 λέγοντας ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ιστορικά στοιχεία και ε, η τροπολογία αυτή ε, είναι, ε, έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο αλλά την αποδέχθησαν και οι Ισπανοί και Πορτογάλοι συνάδελφοι αλλά σε αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, για να ξεκινήσω να σας ευχαριστήσω όλους, όλους όσοι βοηθήσατε για την έκθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε, οι σκιώδεις συγκητές, αλλά και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Αλίας. Καταλήξαμε ε, σε ευρεία συνένεση και ψηφίσαμε την έκθεση με αποτέλεσμα την ε, ομοφωνία για τα οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο στόχος μας είναι να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα ΤΑΚ στη Βαλτική και να σταματήσουμε τις ε, απορρίψεις ε, αλλά και τον λανθασμένο υπολογισμό των ΤΑΚ διότι ε, κάποια πράγματα πρέπει να ισχύουν για ορισμένα μόνο είδη ψαριών. Πάρα πολύ σημαντικό, το άρθρο 15α του κανονισμού 2087 του 87. Το παραλίευμα δεν είναι συνήθως κάτι το οποίο τρώγεται και άρα θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την απόρριψη ζώντων ε, ψαριών που δεν έχουν εμπορική αξία. Επομένω, το εν λόγω άρθρο το 15α θέλει να μα οδηγήσει σε βιώσιμη διαχείριση των ελευτικών πόρων και θαλασσίων πόρων. Επομένω, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη ρύθμιση στη Βαλτική θάλασσα, διότι πολλέ φορέ θα πρέπει να επιβάλλουμε απόλυτη απαγόρευση τέτοιου είδου απόρριψη. Και έτσι να μπορέσουμε να ε, πετύχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση των ε, θαλασσίων πόρων. Πάντω, εάν έχουμε απόλυτη ε, απαγόρευσε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται ούτε για το καλκάνι ούτε για άλλα ε, ψάρια. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το απόθυμο που υπάρχει και προσοχή επομένω γιατί μία απαγόρευση 100% θα αποτελεί μόνο μία πρόφαση για να νομιμοποιηθεί ε, κάποιο είδους μαζική αλίευση βακαλάου, ο οποίος όμως δεν έχει το προβλεπόμενο μέγεθος και είναι μικρότερος. Άρα θα πρέπει τώρα να κάτσουμε και να καταγράψουμε προσοχή τι γίνεται με τα αλίευματα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται ε, τα αλίευτικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος 100% ε, των ε, αλλιευμάτων που εκφορτώνονται και μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια μακρόπνοη πολιτική η οποία να πιάνει τόπο και έτσι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει επομένω να υπάρξει νομοθετική πλαισίωση της αλίας στην Βαλτική. Προσοχή όσον αφορά τους βιομηχανικούς τρόπους αλίας ε, γιατί είναι αλήθεια ότι η Βαλτική ε, είναι ευαίσθητη από πλευράς περιβαλλοντική. ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή ονομάζεται και ε, έχει ένα οικοσύστημα πάρα πολύ ευαίσθητο. Είναι από τα πιο ευαίσθητα στον κόσμο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές διότι τα ψάρια τείνουν να προσαρμόζονται, τείνουν όμως και να μεταναστεύουν, τείνουν να αλλάξουν τις περιοχές όπου ε, γεννούν, στους τόπους οτοκίας και θα πρέπει μέσα να γίνει μια αναφέρωση προστατευμένων περιοχών της Βαλτικής θάλασσας και να υπάρξει κάποιος μακρόπνοη ε, πρόβλεψη για τα καλκάνια. Έχουμε κάποιες περιοχές οι οποίες ε, εξαιρούνται της προστασίας, όμως θα πρέπει τις μεταβολές να τις λάβουμε υπόψη, να προσαρμοστούμε και να δούμε τι θα γίνει με τις προστατευόμενες περιοχές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εισαγωγή των ξενικών ειδών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία διαταραχή των οικοσυστημάτων και ένα από τα βασικά, ένας από τους βασικούς λόγους απώλειας της ε, βιοποικιλότητας παγκοσμίω. Όπως γνωρίζει η Επίτροπος, η εισαγωγή στις παράκτης περιοχές των ξενικών ειδών ε, στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει μέσω πολύ σοβαρών και αυστηρών κανόνων. Ο κανονισμός της Επιτροπής για τη χρήση της διδατοκαλλιέργειας ξενικών ειδών ή απόντων ειδών θα πρέπει να ε, προκύπτει από πορίσματα ερευνών και να μην ξεχνάμε τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, το έργο ΙΜΠΑΣ που μετράει στο, τον αντίκτυπο των, ε, της εισαγωγής τέτοιων ειδών στο περιβάλλον. Εκεί σε κλειστές εγκαταστάσεις έχουμε λεπτομερή αποτελέσματα για τις συνέπειες που προκύπτουν από την εισαγωγή και η, περιγραφή του προγράμματος καθώς και οι λεπτομέρειές του δείχνουν ότι μπορεί σε παραδεκτά επίπεδα να μειωθεί ο κίνδυνος από την εισαγωγή ε, ξενικών ειδών και να αποσβεστεί και ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από τις ε, διαρροές στην ε, μεταφορά, ώστε να είναι ασφαλείς οι εγκαταστάσεις αυτές. Βάσει των αποτελεσμάτων λοιπόν του έργου αυτού, η Επιτροπή προτείνει διευκολύνσεις περιτές δηλαδή για την αδειοδότηση και την εισαγωγή και τη μεταφορά των ειδών αυτών, των κλειστών εγκαταστάσεων, στις κλειστέ εγκαταστάσεις, προτείνονται κανόνες που δεν είναι κατάλληλοι. Αν λοιπόν η διαδικασία της αποτίμησης του κινδύνου δεν βασίζεται σε επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και συμπεράσματα, τότε είναι πολιτική σημασία πλέον το θέμα για το αν μπορούμε να αποδεχτούμε τον κίνδυνο που προκύπτει. Η διευκόλυνση εισαγωγή ξενικών ειδών στι υδατοκαλλιέργειε θα πρέπει να έχει ω αντίβαρο έναν ορισμό πιο αυστηρό ε, όσο δυνατόν των προποθέσεων για τι κλειστέ ε, καταστάσει υδατοκαλλιέργεια βάσει και των απορισμάτων του έργου ΙΜΠΑ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να επιβληθεί φορολογία στι εγκαταστάσει ώστε όλε οι απαιτούμενε τεχνικέ, ε, οι απαιτούμενοι όροι όπως τους θέτουν οι εμπειρογνώμονε, γίνονται σεβαστοί για να λειτουργεί σωστά η κάθε εγκατάσταση. Και επίσης για τη μεταφορά των, ε, ε, των ειδών αυτών είναι σημαντική για το πώς θα λειτουργούν οι εγκαταστάσει αυτές. Γι' αυτό όλα τα στοιχεία αυτά θα τα λάβουμε υπόψη στην σύνταξη της νομοδότησης και θα κάνουμε και τροπολογίες φυσικά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Και μια πρόσθετη παρατήρηση. Η βιώσιμη ε, καλλιέργεια της ε, πολιτικής αλίας πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική και τεχνική γνώση για τους αυτόχθονες ε, οργανισμούς ε, ώστε να υπάρχει διατροφική ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ε, στα ψάρια και να έχουμε βεβαίω ε, και περιβαλλοντική ισορροπία. Η κάθε νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν στον τομέα αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία του τομέα. Πρέπει βεβαίω να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε τη αλληλευτική πολιτική όμως υπάρχουν και δυνατότητες βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να τεθεί σε... πρέπει να αξιοποιηθεί στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Θα ευχαριστήσω λοιπόν εδώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύτιμη συνεργασία τους, την επικοδομητική συνεισφορά τους, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου ε, που και από την Ισπανική Προεδρία αλλά και τώρα με τη Βελγική Προεδρία μας βοήθησαν σε όλο το έργο αυτό που είχαμε να επιτελέσουμε τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ. Κυρία Δαμανάκη, έχει το λόγο. Ε, dear Mr. President, members. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Να πω δύο λόγια για το προολιετές πρόγραμμα για τον Γάβρο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια, την κυρία Μπιλμπάου και όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλίας για το έργο τους στην πρόταση αυτή. Θα ήθελα να πω στην κυρία Μπιλμπάου ότι πράγματι υπήρξε καθυστέρηση. Δεν υιοθετήθηκε γέρος η πρόταση αυτή. Όμως πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά σαφέ ότι η Επιτροπή έκανε ό,τι περνούσε το χέρι τη πραγματικά τα πάντα για να απομπλέξει, να την κατάσταση αυτή. Το απόθεμα γάβρου στον Βυσκαϊκό κόλπο ε, δεχόταν πολλέ απειλέ και είχε πάψει η λήψη νέων αλληλευτικών μέτρων από το 2005. Ξανά άνοιξε τον Ιανουάριο του 2010, ωστόσο. Και τον περασμένο Ιούλιο οι επιστήμονε διαβεβαίωσαν ότι απόθωμα ήταν απάνω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Κάτι που μου επέτρεψε να προτείνω μια ποσόστοση τάκ πάνω από 50.000 τόνους, αυτό που και τώρα ισχύει. Η ποσόστοση αυτή βασίζεται στους αυστηρότερους κανόνες του ε, προγράμματος και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι η πρόταση αυτή ήδη μας εξυπηρετεί στο να διαχειριστούμε ε, επαρκώς το απόθεμα. Αυτή η μακροπρόθεσμη πάυση είχε πλήξει οικονομικά όσους εξαρτώνται από αυτού του είδους την αλληλεία. Πρέπει λοιπόν αυτό να το παρεμποδίσουμε στο μέλλον, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξαναγίνει. Ο μόνος τρόπος που να το κάνουμε αυτό είναι να αξιοποιήσουμε το απόθεμα ε, με βάση την ε, μακροπολιετή αποτελεσματική σοδιά αλλά και με εντατική παρακολούθηση της αλληλευτικής εξέλιξης εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό μπορεί να γίνει αν την ίδια στιγμή παρέχουμε και βιωσιμότητα στην αρμόδια βιομηχανία. Αν Θέλουμε λοιπόν να, πάψουμε, να αντιμετωπίσουμε την πάψη της ε, αλίας, θα μπορούσαμε να βασιστούμε το ποσοστό του 30%. Να ευχαριστήσω εδώ λοιπόν, την Επιτροπή Αλίας και για την επί της ουσίας βοήθειά της, αλλά και για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς την Επιτροπή. Εδώ μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες αυτές και πρέπει να πω ότι θα συμφωνήσω και με τις τροπολογίες που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση της πρότασης με νέο κανονισμό, τον νέο ελεκτικό κανονισμό που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2010. Υπάρχει μόνο μία εξαίρεση εδώ παρόλα αυτά, η οποία έχει να κάνει με τη μείωση, τον περιορισμό της καθυστέρησης για την ενημέρωση ε, ε, ελιμενισμού από 14 σε 1 ώρες. από 4 μάλλον σε μία ώρες. Αυτό προβλέπεται από τον ελεκτικό κανονισμό που ισχύει πλέον. Ξέρετε ότι ο νέος αυτός κανονισμός ισχύει. Ισχύει από την αρχή της φετινής χρονιάς. Έχει τεθεί σε ισχύ και δεν θέλω τόσο γρήγορα να περάσουμε σε τροποποίησή του. Ιδίω επειδή ο κανονισμό για το σύστημα ελέγχου ο ίδιο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ειδικέ εξαιρέσει και ειδικά μέτρα όταν αυτέ δικαιολογούνται. Οπότε είναι κάτι που καλύπτεται. Δεν υπάρχει λόγο να αλλάξει αυτό ο κανονισμό τόσο γρήγορα. Βεβαίω, από εκεί και πέρα επαφίεται σε εσά το θέμα. Τώρα να ε, γυρίσω στην δεύτερη ε, έκθεση, το να στραφώ μάλλον στη δεύτερη έκθεση, το πολιτέ σχέδιο για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού. Ε, ο κύριος Γκάλαχερ έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο μαζί με το μέλη της Επιτροπής Αλίας και να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και για τις σκληρές σας προσπάθειες και για την επικοδομητική σας προσέγγιση. Για το Σαφρίδι πρέπει να πούμε ότι βεβαίως το απόθεμα αυτό είναι το σημαντικότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι σταθερό σε καλά επίπεδα και μεταφράζεται σε σχεδόν αμετάβλητα ποσοστώσεις για το 2011. Η ετήσια απόφαση για το ΤΑΚ, την ποσόστοση για το είδος αυτό, βασίστηκε σε επιστημονικές γνώσεις. Και Βεβαίως θέλουμε να έχουμε μια πολιτική και δεσμευτική προσέγγιση διαχείρισης. Άρα το σχέδιο αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ξεφύγουμε από τα πολιετή πλαίσια του Συμβουλίου για το πόση αλληλεία μπορούμε να έχουμε. Θέλουμε να επιτρέψουμε στη βιομηχανία περισσότερη δυνατότητα προγραμματισμού και σταθερότητα, συμφωνώντα σε πολιετή πιο διορετικά σχέδια, γενική σα στήριξη και στι συγκεκριμένε λεπτομέρειε και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων δείχνουν ότι έχουμε κοινού στόχου. Μπορώ λοιπόν να στηρίξω και τι τροπολογίε σα και αυτέ που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση τη πρόταση με το νέο κανονισμό ελέγχου που ισχύει, όπω είπα, από τον Ιανουάριο του 2010. Πέραν αυτού, το ίδιο το σχέδιο δεν θα πρέπει να αφήσει ακάλυπτες κάποιες περιοχές τάκ ή να μεταβάλλονται αιτήσει αποφάσει ΤΑΚ ανάλογα με τι κειμενόμενε επιστημονικέ συμβουλέ. Υπάρχει ωστόσο μια τροπολογία η οποία δεν οδεύει πιστεύω προ τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα το ότι αποδέχεστε την ε, συμβιβαστική λύση τη Προεδρία του Συμβουλίου για συν ή πλην 5.000 τόνους. Ο αριθμός αυτός, 5.000 τόνοι, είναι αβάσιμος επιστημονικά. Πώς θα αποφασίζουμε εάν θα είναι 5.000. Γιατί να μην είναι 6-7.000. Ε, η διακριτική ευχέρεια λοιπόν να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τα επίπεδα των ΤΑΚ σε ένα πολιετέ ε, πρόγραμμα, μια πολιετή στρατηγική, δεν μου φαίνεται ε, λογική προσέγγιση. Και τώρα να στραφώ στην τρίτη έκθεση για τα μέτρα για τη Χωματίδα και το Καλκάνι στη Βαλτική. Εδώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Γκρομπάρτσικ, για το ε, σκληρό του έργο και για την έκθεση που κατάφερε να εγκριθεί ομόφωνα. Και εδώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αλία για την ε, συνεισφορά τη. Με την πρόταση αυτή βεβαιωνόμαστε για την νομική συνέχεια τη πολιτική μα και ότι θα έχουμε συνέχεια στα μέτρα που άρχισαν να ισχύουν στη Βαλτική από πέρυσι. Ειδικά για κάποια είδη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τώρα να επικεντρωθώ στην τελευταία έκθεση που συζητάμε σήμερα για την χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απότων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Εδώ να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, τον κύριο Φερέιρα, για το έργο του και την Επιτροπή Αλίας συνολικά. Όπω θα ξέρετε, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει ε, την βιώσιμη ανάπτυξη τη αυτοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συγκεκριμένη στρατηγική για την αυτοκαλλιέργεια. Αυτό σημαίνει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντική προστασία αλλά και την θέσπιση προϋποθέσεων και όρων ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Το χρειαζόμαστε αυτό. Η σημερινή τροποποίηση του κανονισμού για την αναπαραγωγή των ξενικών και απόντων ε, ε, σε τοπικό επίπεδο ειδών και την εισαγωγή τους σε ε, καταστάσεις υδατοκαλλιέργειας θα διευκολύνει άροντα, έροντας το διοικητικό άχθος ενώ θα διασφαλίζει ταυτόχρονα πρόσθετη προστασία στα υδάτινα οικοσυστήματα όμω, αυτό δεν είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και καλωσορίζω την πρόταση του κυρίου Φερέιρα να ενισχύσουμε τι ερευνητικέ μα προσπάθειε στην εδωκαλλιέργεια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσω των πόρων του προπολογισμού αλλά και της ανασχετικής μεταρρύθμισης. Χαίρομαι ιδιαίτερος που η συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας κατέληξε σε καλύτερο ορισμό των κλειστών εγκαταστάσεων αντιτοκαλλιέργεια. Να τονίσω εδώ ότι η αρχική πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή ένα μήνα πριν την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα διότι η Επιτροπή Αλίας πρότεινε τροπολογίες που θέλουν ε, να ευθυγραμμίσουν τον νέο κανονισμό ε, με, τους κανόνες περί επιτροπολογίας της νέας συνθήκης. Η ευθυγράμμιση αυτή που προτείνεται από το Ευρωκοινοβούλιο είναι λογική. Έπρεπε όμως και επισήμως να τροποποιηθεί η δική μας πρόταση ώστε να καλυφθούν τέτοιε ουσιαστικέ διορθώσει. Γι' αυτό και προέκυψε σχετική καθυστέρηση. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητέ και τα μέλη της Επιτροπής Αλίας για τις εκθέσεις τους και για το έργο τους σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχουν ομιλητές εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ε, πρώτη η κυρία Φράγκα Στέβες, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τους επιμέρους εισηγητές γιατί ήταν τιτάνιο το έργο το οποίο επετέλεσαν. Θα ήθελα να σας πω τώρα για τα προγράμματα ε, διαχείρισης αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα ουσίας όπως τα ανέδειξαν ε, και οι εισηγητές. Όμως θα πρέπει να σας πω και για τις διάφορες θεσμικές προκλήσεις που έχουν αναδειθεί και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε το Κοινοβούλιο με υπεύθυνο τρόπο και μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο εξέτασε σε πρώτη ανάγνωση αυτές τις εκθέσεις και θεωρήθηκε ότι έτσι θα ασκηθεί μια πίεση και θα απεμπλακεί η κατάσταση διότι έτσι επηρεάζονται και αυτές οι προτάσεις αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια εξέλιξη των προγραμμάτων για το άμεσο μέλλον και εμεί αναζητούμε μια ε, συμβαστική λύση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Για να το πετύχουμε όμω, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι βασικά το Συμβούλιο να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ότι η καρδιά αυτών των προγραμμάτων διαχείρισης μακρόπνο είναι ε, το να υπάρξει κάποιο είδους νομική βάση η οποία να είναι το άρθρο 43 παραγραφός 2 και θα πρέπει δυνάμει τη Λισαβόνα, δυνάμει αυτών των αποκλειστικών ε, αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου για ποσοστώσει και τάκ να γίνεται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Και επομένω θα πρέπει το Συμβούλιο να κάνει αυτά το οποίο επιτάσσουν όλοι οι νομικοί, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνεται περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 43 παράγραφος 2. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, αν μπορείτε απαντήσετε στην κυρία Μπιλμπάου, κατά πόσον κάποια από αυτές τις προτάσεις αντικαταστάθηκε, αποσύρθηκε, αν είχαμε νέα κείμενα. Ε, έχετε την θέση του Κοινοβουλίου, όμως ε, αν συγχθεί έτσι η κατάσταση θα πρέπει να προσφύγουμε ή στο δικαστήριο για να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε την κατάσταση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το επιθυμητό, μια που πρόκειται για ένα πάρα πολύ πολύτιμο εργαλείο για τον κλάδο της αλίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Δαμανάκη. Είναι πάρα πολλέ οι τεχνικέ λεπτομέρειε που έχουν αυτά τα κείμενα που συζητάμε σήμερα. Όμω πίσω από τι τεχνικέ λεπτομέρειε υπάρχει μια ξεκάθαρη εντολή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από του υπόλοιπου θεσμού την Επιτροπή και το Συμβούλιο, οποτεδήποτε αποφασίζουμε για τα θέματά μας το πόσο αλλιεύουμε να σεβόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα. δεν είναι δυνατόν όταν αποφασίζουμε για το πώ θα αλλιεύσουμε κάθε είδος ε, αλίας, κάθε, κάθε είδος ψαριού να διαπραγματευόμαστε με πολιτικό τρόπο. Να υπάρχει μια πολιτική διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο είτε στο Κοινοβούλιο για πράγματα που πρέπει να κριθούν ε, με επιστημονικά δεδομένα μόνο με τα βάση τα επιστημονικά δεδομένα μπορούμε να γνωρίζουμε τι περισσεύει από τις θάλασσές μας τι μπορούμε να αλλιεύσουμε να ψαρέψουμε χωρίς να υπάρχουν ε, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο για τη ζωή στη θάλασσα όσο και για την αλλία. Μπροστά μας έχουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αυτό που σας ζητάμε με αυτές τις εκθέσεις είναι να προβείτε τολμηρά να προχωρήσετε τολμηρά στη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής σεβόμενοι ακριβώς αυτή την αρχή το σεβασμό στα επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να λαμβάνουμε αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις θάλασσές μας και την αλία. Ευχαριστώ πολύ. Ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι θα ε, επικεντρώσω την προσοχή μου στην έκθεση για τον Βυσκαϊκό. Έχω ορισμένε απόψεις επί του θέματος, διότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευαίσθητης ε, των ε, ε, ευαισθήτων ε, ειδών αλληλείας. Είδαμε το 2005 κατέρευσε η αλληλεία αυτή και τώρα είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ σωστά. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτή είναι η άποψη της πολιτικής μου ομάδος. Πιστεύω ότι ο κλάδος της αλληλείας θεωρεί Ε, ότι καλύτερα να λύσουμε τα προβλήματα τώρα παρά να τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Η κυρία Λέμπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει τις εξουσίες του Κοινοβουλίου στα θέματα της αλληλείας και εδώ είναι η πρώτη δοκιμασία για το πώς ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει πολύ καλά, αλλά θεωρήσαμε ότι περάσαμε και δύσκολες στιγμές. Δεν μπορεί κανείς να συμβιβάζεται σε θέματα επιστημονικών συμβουλών διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους αλλοίς αλλά είδαμε ότι η υπεραλληλία οδήγησε σε κατάρρευση και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη των αποθεμάτων και καλύτερα είναι να είμαστε προληπτικοί παρά ε, να παίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε πώς αναπτύσσονται τα ίδια αυτά όπως ε, το είχαμε δει και σε μία ταινία The End of the Line αλλά και εκεί ο σκηνοθέτης είπε ότι υπήρχε ένας αστάθμητος παράγων και αυτός πρέπει να ληφθεί υπόψη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρξει υπέρτατη αξιοποίηση των αλληλευτικών πόρων σε πέντε χρόνια και δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευόμαστε όλα τα είδη συγχρόνως θα πρέπει να υπάρχει ένα, ένα περιθώριο ασφαλείας και ένα όριο όχι δηλαδή στόχος υπεραλίας και ελπίζω ότι έτσι θα διαμορφωθεί στο μέλλον η αληφτική μας πολιτική και θα ε, γίνει αυτό σε συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προστατεύσουμε τα οικολογικά συστήματα της Ευρώπης και όπως είπε και ο κύριος Γκάλαχερ πολύ σωστά το ε, σαφρίδι δεν πρέπει να υπεραλλιεύεται γιατί είναι ενάντια στις απόψεις των επιστημόνων. Τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ είναι θέματα που αναφέρονται και εις το Βόρειο Θάλασσα ή στην περιοχή μου συνάντησα άλλη στην περασμένη εβδομάδα η οποία ανησύχησαν για τα αλλιευτικά σκάφη ή στον Βρετανικό στόλο διότι οι μέρες μειώθηκαν από 135 για την αλληλεία στις 90. Ε, μπορεί ίσως ε, το ποσοστό αυτό της μειώσεως να τους οδηγήσει στη χρεοκοπία και γι' αυτό ανησυχούν. Ε, θα ε, πρέπει βέβαια να λάβει κανείς υπόψη και τις απορρίψεις Δε, όσα ψάρια είναι ζωντανά πρέπει να αποβιβάζονται θα πρέπει να κρατήσουμε το σύστημα διότι η αναθεώρησή του μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του για να μην υπάρχει μία κρίση ποσοστώσεων και η κερδοσκοπία πρέπει να σταματήσει τελείως. Σας ευχαριστώ. Τώρα στους υπόλοιπους εγγραμμένους ομιλητές, ο κύριος Ράγκελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητέ συνάδελφοι. Σε σχέση με την έκθεση Γκάλακερ και ιδίω για, το για το πρόγραμμα διαχείρισης και για το τι γίνεται με το σαφρίδι, είναι καθοριστική σημασία να λάβουμε υπόψη σχετικά την τροπολογία του ΕΛΚ η οποία είναι, συντάχθηκε από το χέρι της ε, συναδέλφου Πέτροβες. Εδώ είναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους τρεις στόχους της πολιτικής αλίας. Τον περιβαλλοντικό που τον γνωρίζουμε όλοι, αλλά και τους οικονομικούς και κοινωνικούς. Πρέπει να υπάρχει οικονομική ωφέλεια, να υπάρχει δυνατότητα επιβίωσης για τους επαγγελματίες του χώρου αυτό. Υπ' αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε την ε, εξόντωση. Μιλάμε για το, απόθεμα, για το δυτικό απόθεμα Σαφριδίου. την ε, περιοχή 8α και στην 8 ε, όμικρον και την περιοχή της ε, του, της Καταβρίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή και της Γαλλίας και της Ισπανίας, αλλά και για την λίγο πιο την περιοχή ελαφρώ περισσότερο στα βόρεια, που είναι σημαντική για τη βιομηχανική αλεία και για την ε, οικονομική επιβίωση. Γι' αυτού λοιπόν του λόγου πρέπει να υπάρξει τροπολογία σε αυτή την έκθεση, ώστε να εραμονιστεί όχι μόνο με του βασικού στόχου τη αλία, τη πολιτική αλεία, για την κοινή πολιτική που θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε δηλαδή, αλλά και με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το, η έκθεση για την προσαρμογή των ποσοστώσεων για το 2011 διότι το σαφρίδι στο ζώνη 8C και στα βόρεια της δυτικής αυτής γεωγραφικής περιοχής που είναι σημαντική για την βιομηχανική αλία πρέπει να ληφθεί μέρημνα. Ε, η τάση αυτής της γεωγραφικής περιοχής είναι να οδηγεί στην εκπλήρωση όλων των στόχων της πολιτικής αλίας ταυτόχρονα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια για τους τέσσερις εισηγητές, για τα προγράμματα διαχείρισης, για τον ε, Γάβρο, αλλά και για το Σαφρίδι χρειάζεται να έχουμε μια βιώσιμη διαχείριση. Ήταν περίπλοκα τα πράγματα και συνεχίζεται η εμπλοκή σε επίπεδο συμβουλίου. Ο κλάδος έχει θυγεί περισσότερο από όλους. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια παράλυση ολοκληρωτική γιατί δεν είχαμε την απεμπλοκή του θέματος γιατί δεν μπόρεσε το Συμβούλιο να λάβει κάποιες αποφάσεις αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να τονίσουμε τους σοσιαλιστές Ισπανούς οι οποίοι σε όλη αυτή τη διαδρομή ε, υπεστήριξαν τα αιτήματα του κλάδου τα ομόφωνα σε σχέση με τα ε, ΤΑΚ για τα όσα έχουμε ζητήσει να καλυφθούν από την μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής. Θα πρέπει να αποσυρθεί μας λέτε η έκφραση και θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις δικές μας θέσεις για μια νέα πρόταση. Τώρα, όσον αφορά το Σαφρίδι, έχουμε αυτά τα ζητήματα που ανέδειξε ο εισηγητής. Εμείς συμφωνούμε με τα όσα ελέγχθησαν για, τη, για πολιτική προγράμματα, για τα ΤΑΚ, για τις εισηγήσει των επιστημόνων. Συμφωνούμε με όλα αυτά και έχουμε μια τροπολογία. Η σοσιαλιστική ομάδα θεωρείται ότι είναι σημαντική και οι Ισπανοί σοσιαλιστές επίσης, μια που στη χώρα μας Έχουμε την παραδοσιακή αελία του σαφριδιού που τη μέρα που ψαρεύεται το, το, ψάρι καταναλώνεται. Όμως προσοχή μήπως με τις νέες ρυθμίσεις έχουμε κοινωνικο-οικονομική ζημία και πλήγματα στον κλάδο και έτσι επομένως θα πρέπει να κάνουμε τις ρυθμίσεις που απαιτεί καλύτερη διαχείριση κύριε Γκάλαχερ παρακαλούμε λάβετε υπόψη την τροπολογία μας όσον αφορά την παράκτη ελία. Για ένα λεπτό.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 Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, λόγω των ε, πολλών εισαγωγών των ψαριών θα πρέπει να προωθήσουμε την υδατοκαλλιέργεια. Χρειαζόμαστε την δυνατότητα και οι αλληλείς μας να έχουν καλύτερη δυνατότητα επιβιώσεως και ε, να έχουμε περισσότερους πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν να, να υπάρξει καλύτερη έρευνα και καλύτερα στοιχεία τι μόνο αν γνωρίζουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει θα μπορέσουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Η, ε, η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη γνώσης είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να συνδυάσουμε την οικονομία και την οικολογία, δύο στοιχεία τα οποία δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενο ομιλητή ο κ. Ρωμέβα Ερουέδα. Για το γάβρο. Θέλω να σα τονίσω το πόσο σημαντική υπόθεση είναι αυτή η ρύθμιση για τον κλάδο αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Είναι ξεκάθαρο το πόσο οι πράσινοι υποστηρίζουμε αυτές τις προτάσεις. Αυτό που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνούμε πρώτα από τα όσον αφορά τον τρόπο εκμετάλλευση. Συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να πάμε, πηγαίνουμε πάνω από το 0,3. Συμφωνούμε επίση με την Κομισιόν για το ΤΑΚ ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντα ζωντανό δόλωμα. Και επίση θα πρέπει να, έχουμε, να φτάνουμε εκεί πέρα μέχρι το 25% όπω προτείνει η Κομισιόν. Θεωρούμε ότι είναι επομένω λογικέ οι προτάσει τη και επομένω θα πρέπει. Ε, ε, επιτέλους για κάποια φορά να ε, δρούμε σαν ένας γιατρός και όχι σαν νεκροτόμος. Κάποιος δηλαδή που να προλαμβάνει το πρόβλημα και μην έρχεται μετά να διαπιστώσει το, το, το, το, πλήγμα που, ε, που δημιουργήθηκε. Κούν δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η δικιά μου συμβολή αναφέρεται εις την απαγόρευση ε, της αλληλείας εις τη Βόρειο Θάλασσα και στο Άρεσουν. και εδώ πρόκειται για δύο συγκεκριμένα θέματα ε, πρόκειται για δύο είδη ψαριού τα οποία χρειαζόμαστε στην αγορά μας και διαπιστώνουμε ότι είναι ανάγκη εδώ η ε, επιστήμη ε, και οι εμπειρογνώμονες να συνεργαστούν κατά τρόπον ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων μας και αυτό να αξιολογηθεί ε, και, και το θέμα της παρεμπίπτωσης των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτά τα θέματα θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό διότι όπως ακούσατε ο εισηγητής είπε πολύ σαφώς και αυτό ήταν ο στόχος μας τον οποίο επιτύχαμε ότι μειώνουμε μεν το, τις απορρίψεις και το παρεμπίπτον αλίευμα αλλά έχουμε και μικρά ψαράκια τα οποία εάν αλλιευτούν μετά μπορούν να ξανααπορριφθούν στη θάλασσα πράγμα το οποίο μπορεί να ε, μας επιτρέψει να κάνουμε επιλεκτική αλία γιατί θα πρέπει ε, να, ε, ε, να διευθυνίσουμε ακριβώς ποιος θα είναι ο χρόνος της αλληλείας να μην τροποποιήσουμε τις παραμέτρους κατά τρόπον ώστε να μην χρησιμοποιούνται εξαιρετικά ψάρια για να δημιουργούνται απλώς ζωοτροφές και χθιάλευρα και γι' αυτό χρειάζεται χρειάζεται να αλλάξουμε το σύστημά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόνταστ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρία Δαμανάκη, χαίρομαι διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε τέσσερις βασικούς κανονισμούς του οποίου θα υιοθετήσουμε για την αλληλεία και θα αναφερθούμε και στην υδατοκαλλιέργεια και στα μέτρα αλληλείας στα οποία συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά στην Επιτροπή μας πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την αξιοποίηση των αποθεμάτων γάβρου. Νομίζω ότι οι προοπτικές για την Ολομέλεια είναι πολύ καλές και ελπίζω ότι εντωμεταξύ άλλαξε γνώμη και ε, το ΕΛΚ που δεν υπέβαλε άλλες τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν ότι και αυτοί ε, θα επικροτήσουν αύριο στην ε, ψηφοφορία. Το πρόβλημα όμω είναι με το Συμβούλιο, διότι η πλειοψηφία των κρατών ε, εν αντιθέσει με τους νομικούς συμβούλους της δεν δέχεται την συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από ένα χρόνο που ισχύει η θήκη της Λισαβόνας και το βρίσκω παράδεκτο. Γι' αυτό και πρότεινα να στείλουμε μια κοινή επιτροπή στους Υπουργούς Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ήθελα εντός των επομένων εβδομάδων να συμφωνήσουμε κατά τρόπον ώστε να δείξουμε ότι κινείται ενιαία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην το καταπιεί το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Χάτστον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα συμφωνήσω με τη γραμμή του κυρίου Γκάλαχερ και τις εκθεσής του και θα ψηφίσω αναλόγω βεβαίως αύριο όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Να πω απλώς ότι η αρχή του πολιετού προγραμματισμού είναι πάρα πολύ λογική. Το θέμα όμω είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δουν σε πολιτή βάση την ε, ζωή του και οι ίδιοι οι ψαράδε. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ αρνητική πτυχή της, ε, του πρόγραμματο διαχείριση ε, τη ελληνική πολιτική στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι γίνεται με τι πωλήσει, με περιοχές που υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ε, αποφάσεις και απαγορεύσεις λόγω των μέτρων διατήρησης των αποθεμάτων. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις απορρίψεις. Υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη δυσφορία σε σχέση με τις απορρίψεις ως αποτέλεσμα των κανόνων των ευρωπαϊκών μέτρων. Επίτροπε, πρέπει να λάβετε δράση για να ασχοληθείτε και με αυτό το μέρος του σκανδάλου των απορρίψεων που είναι κάτι που προκύπτει από τους ισχύοντες κανονισμούς και μας επιβαρύνει ιδιαίτερος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάτο Αντρόβερ για δύο λεπτά θέλω να μιλήσω για δύο από τις εκθέσεις που νομίζω ότι αποτελούν παράδειγμα μίμησης και αποφυγής για το γάβρο αλλά και για την εκτιοκαλλιέργεια και τα εξωτικά είδη για τη γάβρο ε, ε, αυτό είναι παράδειγμα προς αποφυγή διότι πάνω από ένα χρόνο μιλάμε και συζητάμε και τελικά η συζήτηση ε, επικεντρώθηκε στο ποιε είναι οι αρμοδιότητες σήμερα με συνήθειες Λισαβόνας για μας και ποιες για την Κομισιόν. Δεν συζητήθηκε το τι είναι καλύτερο για τους αλείς, για τον κλάδο, για το, το, στόλο. Επομένως το θύμα όλες αυτές τις υπόθεσεις είναι ο κλάδος που ε, με έκπληξη διαπιστώνει το, πώς διεκπεριώνουμε αυτά τα θέματα του και πώς δεν τους βοηθούμε για να έχουν ένα μέλλον. Επομένως, δίκαια παραπονούνται για τις διοικητικούς φραγμούς της πρόοδου για την υπόθεση αυτή. Θέλω να προχωρήσουμε χωρίς ε, τέτοιου είδους ε, διακοπές. Ε, επομένως θα πρέπει και σήμερα να αρθεί αυτή η βεβαιότητα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να στείλει ένα θετικό μήνυμα. Απ' την άλλη μεριά, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι συμφωνήσαμε όσον αφορά αυτά τα εξωτικά είδη σε πρώτη ανάγνωση. Βρέθηκε ο συμβασμό. Τα τρία θεσμικά όργανα ταχαίω τα βρήκανε. Δεν είχαμε ούτε επί ούτε επί των θεμάτων διαφωνία και επομένως τώρα έχουμε τους σωστούς ε, ορισμούς και επίσης έχουμε την ε, ασφαλεία δικαίου που είναι αυτό το οποίο ο κλάδος και επίσης κατά αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να μειώσουμε την ε, γραφειοκρατία που βασανίζει τον κόσμο. Είμαι δε ότι θα πρέπει οι διοικητικέ διαδικασίες να συρρυκνωθούν όσο γίνεται περισσότερο, ούτω ώστε να μην ε, βασανίζεται τόσο πολύ ο Ευρωπαίος για οποιαδήποτε δραστηριότητα που τη δυσκολεύει η γραφειοκρατία. Επομένως, οι διαδικασίες όποτε προβλέπονται είναι κακά μαντάτα για τον κλάδο ε, για να συνεχίσει, ο συνεχίσει φραγμό στην δραστηριότητα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητή, είναι ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Δαμανάκη. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις εκθέσεις Φεραίρα και Γκρόμπατσεκ. Συγχαρητήρια εις τους συγκητές γιατί κατέφεραν ε, να κλείσουν αυτούς τους δύο κανονισμούς που ε, υλοποιούν την συνθήκη της Λισαβόνας για την λευτή δραστηριότητα και έτσι μπορούμε τώρα να έχουμε διαχείριση βιώσιμη όσον αφορά την βιοπικιλότητα. Και επομένως τώρα έχουμε ε, τις ρυθμίσεις αυτές για ε, το, το καλκάνι στην Βαλτική αλλά και, το, και για τα άλλα είδη της ε, Μεσογείου για να μπορέσουμε να έχουμε και στη Μεσόγειο και στη Βαλτική ρυθμίσεις ούτω ώστε τώρα πια σε αυτά τα κοινωτικά ύδατα να, να, να αλλάξει στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ελληνικής πολιτικής η πολιτική που αφορά ε, τις, ε, τις απορρίψεις ε, και επίσης θέλουμε να υπάρχει μια σχετική λίστα η οποία είναι δημόσια να μπορούμε να έχουμε κάποιο, κάποια νομοθεσία που να, να βοηθά το οικοσύστημα και έτσι να μην έχουμε μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο κύριος Καντέκτορ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ του συναδέλφου Μπιλμπάου, Γκάλαχερ, Γκρομπάτζικ και Φεραίρα για τι εκθέσει του. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί βλέπω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ολοκληρώνεται το γύρο τη πρώτη ανάγνωση για δύο πολυετή πρόγραμμα. Για το Σαφρίδι και το Γάβρο. Από την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο ε, συναποφασίζει για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι η Επιτροπή Αλία στοχεύει σε μια πολυετή πολιτική και ένα πολυετέ πρόγραμμα διαχείριση, ώστε να υπάρχουν κοινοί στόχοι για τι χώρε που ψαρεύουν. Έτσι, στις ποσοστώσει λαμβάνονται υπόψη επιστημονικά στοιχεία ώστε δικαιότερα να ορίζονται οι ποσότητες, οι ποσοστώσεις που μπορούν να αλληλευθούν για τα αλλιεύματα, για το σύστημα ελέγχου που πρέπει να είναι κοινό μεταξύ κρατών μελών που εκμεταλλεύονται τα ίδια αποθέματα. Όλα αυτά είναι καθοριστική σημασία για την έκθεση του κ. Γκάλαχερ, τον οποίο συγχαίρω. Ελπίζω αύριο να υιοθετήσουμε μια έκθεση που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση του δυτικού αποθέματο Αφριδίου και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε επίπεδο αηφορία. Γιατί έτσι θα έχουμε ένα σύνολο επιτρεπτών ορίων αλλίευση για σωστή διαχείριση και χρηστή διαχείριση του αποθέματο μακροπρόθεσμα. Να θυμίσω εδώ τη σημασία του, της έννοιας της σχετικής σταθερότητας, την οποία τη θεωρώ πολύ σημαντική. Ο εισηγητής ε, μιλά για την ανάγκη καταπολέμησης των απορρίψεων και συμφωνώ με αυτό. Όμως ε, λυπάμαι που βλέπω ότι το Συμβούλιο ε, αμφισβητεί την νέα εξουσία του συναποφασίζει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιετή πολιτική. Θα πρέπει αυτό το πρόβλημα πολυδυναμικής βάσης να επιληθεί, διότι θα πρέπει για τα προγράμματα που θα τεθούν σε ισχύ να είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε την ε, επιβίωση των αποθεμάτων και το μέλλον της αλίας. Επίσης η ε, βιομηχανική αλία αλλά και η σε μικρότερη κλίμακα είναι σημαντικό να διατηρηθούν ώστε να μεταρρυθμιστεί σε βάση, σε σωστές και γερέ βάσει ε, η πολιτική αλεία. Και εδώ ευχαριστώ τον κύριο Γκάλαχερ για τι προσπάθειέ του. Τώρα, για προγράμματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά, ε, ξέρουμε ότι δεν έχει νόημα να τα επιδιώκουμε. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πρόγραμμα που να δίνει κίνητρα στου εργαζόμενου σε αυτό το τομέα, αλλά να επιτρέπει και οικονομικό όφελο και περιβαλλοντικά κέρδη. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκάλαχερ. Ο κύριο Μιλάνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι λίγη, λίγο ένα λεπτό για να σχολιάσω τέσσερι εκθέσει, αλλά θα σταθώ σε αυτή του κυρίου Φερέιρα. Για την βιοπικιλότητα πρέπει να γίνει επιτακτική ανάγκη η προστασία τη. Ε, όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω ε, εγκρίνει νομοθετήματα για την φωτοκαλλιέργεια και την ελευθερική πολιτική. Η έκθεση του κυρίου Φερέιρα νομίζω ότι καλύπτει τι περισσότερε από τι ανησυχίε μα δεν χρειάζεται να είναι κανείς προκατελημένος κατά της έρευνας ε, και πρέπει σίγουρα να βελτιωθούν τα πρότυπα της αλίας όμως, να είμαστε πολύ αυστηροί και στους ελέγχους και στην οθέτηση προδιαγραφών ώστε να είμαστε ακριβείς στην περιγραφή τους και να αποφύγουμε κινδύνους ε, για την αλλίωση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Εδώ θέλουμε την πρόθεση της βιοποικιλότητας αλλά και να εξασφαλίσουμε προστασία να δίνουμε εγγυήσει και να αξιοποιούμε την, την παραγωγή των αυτοχθόνων ειδών. Κυρία Επίτροπε, όταν βλέπει κανεί τι εξελίξει στην πρωτοκαλλιέργεια, ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν σεβαστά στην ευρεία μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο και απλουστευμένο κανονισμό. Αυτό πραγματικά είναι μια έντονη ευχή μου και ελπίζω να μπορέσετε με το έργο σα να απλοποιήσετε όλε τι διαδικασίε. Ευχαριστούμε και τώρα η διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Είναι αρκετοί ομιλητέ. Ο κύριο Λουέντσα. Για ένα λεπτό. Πρόσε πάνε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από πλευρά μου του συναδέλφου, ιδίω τον κύριο Γκρομπάτσικ, για τη συνεργασία που είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που καλύπτει η έκθεσή του. Ε, και η Επιτροπή εδώ καλείται να εξεύρει ένα συνολικό ένα σφαιρικό πρόγραμμα για την χωματίδα και το καλκάνι στην Βαλτική θάλασσα. Εδώ οι αρχές της Πολωνίας επί πολλά χρόνια συνηγορούσαν υπέρ της ανάγκης συνολικής διαχείρισης του αποθέματος του Καλκανιού στην Βαλτική. Αλλά δεν υπήρχε απόκριση για πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα βλέπουμε ότι χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης για τα ίδια αυτά σε όλους τους οικοτόπους τους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη Βαλτική θάλασσα και τους ψαράδες της, τους πολωνούς ψαράδες. Ε, έτσι λοιπόν το πρόβλημα θα, είναι πολύ καλό που πλέον το έχει λάβει υπόψη της η Επιτροπή. Ο κύριος Κράουλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές και για τις εκθέσεις τους και ιδίως τον κύριο Γκάλακερ. Δύο πράγματα που σκέφτηκα κατευθείαν όταν άκουγα τη συζήτηση που έγινε εδώ. Πρώτα απ' όλα ότι η όλη περιοχή θα πρέπει να δώσει ευκαιρία στον κόσμο της Αλίας μέσω τον ΤΑΚ, αλλά είναι πρόβλημα ευθύνη αυτό που θα πρέπει να αναλυφθεί. Και εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις απορρίψεις. Ίσως πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, όρια. Υπάρχουν παραλιεύματα τα οποία πολλέ φορέ πετιούνται ξανά στη θάλασσα. Γιατί μερικέ φορέ να μην εκφορτώνονται και να καλύπτουν το κόστο των αλλιευμάτων, όχι στην τιμή τη αγορά, στην τιμή τη αλλίευση. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει εκατοντάδε τόνου ε, για την ε, εκμετάλλευση ειδών, την εξαγωγή και εισαγωγή του και να ενισχύσει την αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κατάσταση αυτή που θα μπορούσε να δώσει ωφέλη σε όλε τι πλευρέ και να προσφέρει και στου ψαράδε μα δυνατότητα να έχουν προϊόντα που πουλιούνται. Ευχαριστούμε κύριε Κράουλη. Ο κύριος Γκρίφιν το ζητεί το λόγο. Στα πίσω έδρα είναι πάρα πολύ καλό πρόεδρε ότι δεν κινδυνεύονται που θέλετε να τα σώσετε και έχουμε όλες αυτές τις προτάσεις σας, συγχαρητήρια, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τόσες πολλές προτάσεις έπεσαν στο παρελθόν ε, και ε, με, τις, με την κοινή αληθική πολιτική είχαμε πάρα πολλά είδη στη Βρετανία που ε, εξαφανίστηκαν οπότε θα πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες και όχι τους ευρωκράτες. Επομένω, θα πρέπει τώρα για τα υπόλοιπα ψάρια που έχουν μείνει να σταματήσουμε αυτές τις απαγορεύσεις ε, να έχουμε όχι απαγορεύσεις απόρριψης αλλά ε, περιορισμό του, του, του, του αλλιεύματος σε σχέση με το τι ε, από αυτά τα οποία ψαρεύονται πάνω σε άνθρωπο ή σε άλλες λύσεις και επομένως θα πρέπει να έχουμε ποσοστώσεις που θα πρέπει να, τη, να είναι ιδιοκτησία των αλλιέων και θα πρέπει επίσης να είναι μεταξύ των αλλιέων και επομένως να μην ε, υπάρχει κάποιο συμφεροντοκρατία. Ε, τώρα τον λόγο ζητεί ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι ειδικό, αλλά προέρχομαι από νησιωτική χώρα και γνωρίζω ότι η Ελία είναι πάρα πολύ σημαντική. και επομένω πάρα πολύ εύστοχα Είναι αυτά τα οποία ελήφθησαν όσον αφορά την άστοχη ρύθμιση κάποιων ποσοστώσεων. Σε πολλά διευθυνούμε τον κύριο Γκαλαχέρ, αλλά αυτό το οποίο είπε για το Σαφρίδι είναι σωστά. Άρα θα πρέπει τώρα να μας απαντήσει η Επιτροπή επί τη βάση τεκμηρίωση επιστημονική. Επίση, γίνεται με τι ε, απορρίψει, γιατί γίνεται και με την δεν Θα πρέπει περισσότερο να το προσέξουμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορούν οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν όλα τα είδη ψαριών. Ο επόμενος. Τελευταίος προσπάθησα να υπολογίσω το κόστος της ε, κοινή ληφτικής πολιτικής στη Βρετανική οικονομία και είναι περίπου 6,3 δισεκατομμύρια το χρόνο συν 7,5 ε, δισεκατομμύρια συν γραφειοκρατία και τα λοιπά 2,2 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο με σύνολο 11,1 δισεκατομμύρια. Η αλληλευτική πολιτική έχει καταστραφεί και ε, από το 1973 έχει καταστραφεί ο κλάδος. Το ανθρώπινο κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί. Ε, το περιβαλλοντολογικό αποτέλεσμα είναι τραγικό διότι χάνονται εκατομμύρια ειδών εις τη Βόρειο Θάλασσα θάλασσα και η λύση θα ήταν να ε, εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, αναβιώσουμε την αλληλευτική μας βιομηχανία. Ευχαριστώ και ο κύριος Κόρτες Λάστρα τελευταίος. το 2005 ε, σταμάτησε η αλληλεία στον κόλπο της Βισκάιας λόγω του προγράμματος αναδιάθρωσης. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια βιώσιμη εκμετάλλευση με ποσοστώσεις βάσει επιστημονικών κριτηρίων. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τον κλάδο, κλάδο που χρειάζεται σταθερότητα. Ζητώ από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή τη και να λάβει υπόψη την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Η Επίτροπος κύριε Δαμανάκη έχει το λόγο. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές και για την συνεισφορά τους. Η συζήτηση ήταν πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Πρώτα, να αντιδράσω στις παρατηρήσεις της κυρίας Φράγκα, εκ μέρους του ΕΛΚ και άλλων μελών για τα θεσμικά προβλήματα που έχουν προκύψει πλέον. Ε, αναφερθήκατε στο νέο περιβάλλον του, το θεσμικό που έχει προκύψει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η θέση σε ισχύ της συνθήκης έχει δημιουργήσει πραγματικά, έχει οδηγήσει στην έναρξη μιας νέας εποχής. Και θα πρέπει πραγματικά να το δεχτούμε αυτό. Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως και στηρίζει την ιδέα το Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα λόγου ό,τι αφορά του κανόνε εσοδεία στα πολιετή προγράμματα διαχείριση. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκε είναι πολύ σαφεί όταν αναφέρονται στο, στο θέμα αυτό. Η θέση λοιπόν αυτή είναι η προκατακτική μα θέση, αλλά όπω ξέρετε υπάρχει αντίδραση από το Συμβούλιο. Αντίδραση διότι κάποια κάτι μέλη αντέδρασαν εντόνω και μάλιστα υπάρχει και γενική αντίδραση σε αυτή την προσέγγιση. Οπότε θα πρέπει να εξεύρουμε κάποια λύση εδώ. Ιδάλω δεν θα μπορούμε να ε, θέσουμε σε εφαρμογή τα πολιετή προγράμματα διαχείριση. Και όπω καταλαβαίνετε, τα προγράμματα αυτά είναι το μέλλον μα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε με τη νέα πολιτική όπω την θέλουμε, όπω θέλουμε να τη διαμορφώσουμε, βασιζόμενοι σε παλιέ πολιτικέ νοοτροπίες. Προκειμένου λοιπόν να απεμπλακεί αυτή η κατάσταση, έχω σκεφτεί ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διέξοδο, ίσω με μια τριμερή συνάντηση. Θα προτείνω στο του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε, προκειμένου να βρούμε μια λύση, να υπάρξει μια συμβαστική λύση, η οποία χρειάζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για όλα τα πολυετή προγράμματα διαχείριση υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα, παρα, ε, καθυστερούν και έχουμε και νέα προγράμματα ε, διαχείρισης για τα πελαγικά είδη λόγω χάρη και για τον Σολομό. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πολυετή προγράμματα. Είναι έτοιμα και περιμένουν, περιμένουν να δοθεί θεσμική λύση σε αυτό το πολύ ευαίσθητο πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, συνεισφορά των υπόλοιπων ομάδων, να καλωσορίσω την Συμβολή του κυρίου Αρσένη, του κυρίου Λέβιν από τις διάφορες ομάδες και να συμφωνήσω μαζί τους ότι χρειαζόμαστε πολυετή προγράμματα διαχείρισης ακριβώς και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Καταλαβαίνω εδώ και θέλω να είμαι πολύ σαφής από αυτού ότι αυτό το απαιτούν και οι ψαράδες μας. Είναι πρόβλημα το τομέα της αλίας μας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα μια συγκεκριμένη κατάσταση. <clears throat> Το πρόγραμμα για τον Γαύρο, το γεγονό ότι έπρεπε να πάψει η Αλία και για πέντε χρόνια, κάποια τέλο πάντων χρόνια, ήταν ένα σαφέ μήνυμα, μια σαφή απόδειξη ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λέγοντα ότι αμελούμε και δεν λαμβάνουμε υπόψη τι επιστημονικέ συμβουλέ. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα, εδώ πρέπει να βρεθεί λύση, μια διέξοδο. Όμω, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή θα είναι μια από τι βασικέ κατευθύνσει που θα ακολουθήσουμε στην αλληλευτική μα πολιτική και στη μεταρρύθμιση τη. Προκειμένου να προχωρήσουμε βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία και να βρούμε έναν τρόπο σε περίπτωση που επιστημονικέ συμβουλέ δεν είναι αρκετά ακριβή, δεν είναι ακριβά, αρκετά σαφή. αν δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, να σας πω ότι η έκθεση του κ. Γκορμπάτσεκ είναι πολύ σημαντική. Τα τεχνικά μέτρα για την αποφυγή της ε, ε, αναβάθμισης είναι πολύ σημαντική για την πολιτική μας. Επίση να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε μία πολιτική για τη χωματίδα και το καλκάνι, όπω είπαμε, και θα το πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις, ωστόσο, πολλοί που σας μίλησαν για τις απορρίψεις, χρειαζόμαστε μια θαραλέα πολιτική, πραγματικά θαραλέα πολιτική. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε να πετάμε ξανά ψάρια στη θάλασσα όταν είναι τόσο πολύτιμα. Δεν έχουμε την οικονομική αυτή δυνατότητα. Μπορεί να ήταν μια λύση όταν είχαμε πολλά ψάρια στα ύδατά μας. Τώρα ωστόσο υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, δεν μπορούμε να πετάμε στη θάλασσα ψάρια. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση και καλωσορίζω ιδιαίτερα προτάσεις όπως ε, της αποζημίωσης των αλλιέων για το κόστος ε, των παραλιευμάτων. Να βρούμε λύσεις, ε, αλλά τούτο πρέπει να γίνει μέσω μεταρρύθμισης πολιτικών, προχωρώντας προς ένα στόχο της κατάργησης των απορρίψεων. Βεβαίω πρέπει να έχουμε υπόψη μα τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση εκείνη. Μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε, για τα προβλήματα της υδατοκαλλιέργειας. Πρέπει να μειώσουμε τα προβλήματα επιβάρυνσης και τα εμπόδια επιβάρυνσης στην ε, υδατοκαλλιέργεια. Συμφωνώ με αυτό. Μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή και άλλους ομιλητές που μίλησαν για το θέμα αυτό. Τι θέλω να σας πω ωστόσο, προσπαθούμε να το πετύχουμε κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της κοινής ελευτικής πολιτικής. Θέλω να επιβεβαιώσω και να επαναλάβω ότι θα ενισχύσουμε τις ε, επιστημονικές έρευνες για τα ήδη υδατοκαλλιέργειες, διότι πράγματι χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε προς μια μαζική παραγωγή τέτοιων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αν θέλουμε η υδατοκαλλιέργεια να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην αλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμεί ευχαριστούμε. Οι συγγητές έχουν το λόγο. Η κυρία Μπιλμπάο πρώτη. Κυρία Πίτροπε, καταρχάς, θα ήθελα να, απαντήσετε με σαφήνεια, να είχατε απαντήσει με σαφήνεια. Η πρόθεσή σας είναι να δεχθείτε τις απόψεις του Συμβουλίου αναγνωρίζοντας και ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποδοχή των αρμοδιοτήτων που δίδει στο Κοινοβούλιο μας η Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Αλληλείας ψήφισε για δεύτερη φορά και δεν ζήτησε από την Επίτροπο να αποσύρει την πρότασή της. Ζητή, ζητούμε να απαντήσει η Επίτροπος αν θα δεχθεί τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσει του Συμβουλίου ή όχι. Ο κλάδος απαιτεί πρόγραμμα. Ήταν υπεύθυνο, δούλεψε για δύο χρόνια με την Επιτροπή και με επιστημονικά Ινστιτούτα για να καθορίσει την πρόταση για τον κανόνα της εκμετάλλευσης. Ένας κλάδος ο οποίος μετά από πέντε χρόνια καθυστερήσεων και διακοπής και μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο κλάδος ζήτησε τη διακοπή μπόρεσε να πάρει, να, να αλλιεύσει 7.000 τόνους πέρυσι που καθορίζει κάθε μέρα την ποσόστοση που πρέπει να λιεύσει για να γίνει αποδοτικότερη η μικρή ποσόστοση που μπορεί να χρησιμοποιήσει και που μονομερός αποφάσισε να τις τους ανακοινώσει η Επιτροπή ότι πρέπει να σταματήσουν, να, να, την Επιτροπή να σταματήσουν διότι ε, ξεπέρασαν τον κλάδο, το, το, το, την ποσόστοση. Είναι ένας κλάδος που ποτέ δεν ξεπέρασε αυτά που του, που ζητούσαμε που ζητά απλά διαφάνεια, που, ζει, που δούλεψε με αυστηρό τρόπο για να έχει αυτό το πρόγραμμα που χρειαζόμαστε τόσο. Η έγκριση του προγράμματος αυτού σημαίνει ότι ε, βγαίνουμε από τις ε, αδιαφανείς πολιτικές αποφάσεις. Αυτό ήταν οι αποφάσει για τις ποσοστώσει και τα τάκ. Με αυτή την αδιαφάνεια ζήσαμε πολλά χρόνια. Ο 21ο αιώνα, ωστόσο, δεν είναι ο αιώνα τη αδιαφάνεια, δεν είναι αυτό που, αξίζει, που αξίζουν οι πολίτε τη αδιαφανεια δεν ειναι αυτο που αξιζει αξιζουν οι πολιτε τη ευρωπη και ένα υπεύθυνο κλάδος. Ευτυχώ η τελευταία έρευνα του βασικου Επιστημονικού Ινστιτούτου του Ράστιεφ έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερος γάβρος ξεπεράσετε το όριό της. Θα ήθελα μια απάντηση σαφέστερη από σας κύριε Επίτροπε πάντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Γκάλεχερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους και τους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Γκάλεχερ, μπορείτε να μιλήσετε πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Ξαναρχίστε το χρονόμετρο, κύριε Πρόεδρε. Λέγω ότι ευχαριστώ την Επίτροπο και του συναδέλφου για τι παρεμβάσει του και τους και ηγητές και το Συμβούλιο και την Επιτροπή και του Συμβούλου στην Επιτροπή και τους δικού μου συμβούλους. Καταλαβαίνω ότι γίνεται η συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο και καταλαβαίνω ότι οι 27 υπουργοί πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα υπερισχύσει η κοινή λογική. Αναφέρομαι στη δυσκολία της Επιτρόπου με το συμπλήν 5.000 τόνους. Είπαμε ότι είναι μια πραγματιστική λύση. Το φάκελο αυτό το συζητάμε εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ για να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τι δυσκολίε. Και στου σοσιαλιστέ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισημία για τη θέση μου σε σχέση με την τροπολογία σα. Και σαφώ ε, θα δώσω τη σύσταση να υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Και όσον αφορά την πρόταση του ΕΛΚ, ε, είπα και στο ΕΛΚ ότι πρέπει να το σκεφτούν και εγώ πολύ προσεκτικά συμπεριέλαβα τι ανησυχίε του στην τροπολογία 7 για το βυσκαϊκό κόλπο και για την αναστεχνική ελεία. και οποιοδήποτε υποστηρίζει κάτι τέτοιο θα πρέπει να θυμάται ότι υπήρχαν πάρα πολλέ εκθέσει στο Κοινοβούλιο και αν υποστηρίξουμε τώρα κάτι το οποίο είναι ασφαλμένο ίσω για να είμαστε συνεπεί θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε κάτι ασφαλμένο και στο μέλλον. Είναι λοιπόν απόλυτα εσφαλμένο. Επιστημονικά δεν είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι επιστημονικά εσφαλμένο να διαχωρίσουμε το ΤΑΚ και αν το κάνουμε τώρα θα χρειαστεί να το κάνουμε και στο μέλλον. Και για τα πολιετή σχέδια είναι ζωτική σημασία να επιτρέψουμε στον τομέα να κάνει τον προγραμματισμό για το μέλλον. Ελπίζω ότι αύριο θα υπερισχύσει η κοινή λογική και ότι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση την οποία να μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλεχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριο Γκλέμπαρσικ, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, ε, ε, του κοιόδης συζητητές, κυρία και Ρόντου, τον κύριο Κούνς και την κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ όλου για τα πολύ θερμά του λόγια για τα καλά λόγια που είπαν για την έκθεσή, του, για την έκθεσή μου. Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα μας δώσει τις ε, κατάλληλες λύσεις και θα μιλήσουμε για το περιφερειακό χαρακτήρα στο επίπεδο που χρειάζεται. Γιατί ο περιφερειακός χαρακτήρας είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην κοινή πολιτική αλληλείας. Αυτό θα μας εγγυηθεί την επιτυχία της μελλοντική πολιτικής αλληλείας. Ο Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε σε απάντηση και να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για το πολιετές πρόγραμμα ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Η τροπολογία και τις απόψεις τη η τροπολογία 7 του εισηγητή δεν ε, εξασφαλίζει την διαφοροποίηση τον την αναγνώριση των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε στόλου. Οι διαστάσεις αυτές ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των ΤΑΚ. Η μικρή τοπική και παράκτη αλία έχει ειδικά χαρακτηριστικά που δημιουργεί και κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ε, ο περιορισμός στην αλία ε, ιδίως, ιδίως για περιοχές όπου χρησιμοποιείται η αλληλεία για την ε, παροχή καθημερινού ψαριού για το τοπικό πληθυσμό δεν είναι το ίδιο με την μαζικής παραγωγή αλληλεία. Τέθηκαν ε, και ορισμένα τεχνικά ζητήματα και δεν συμφωνώ με την άποψη του, του εισηγητή. Μιλάμε για το ίδιο στόκ, για το ίδιο απόθεμα, για την ίδια ελία που εξελίσσεται διαφορετικά σε διαφορετικές ζώνες. Η παράκτια και βιοτεχνική αλληλεία δουλεύει σε, συγκεκριμένο, συγκεκριμένη περιοχή, ενώ η βιομηχανική αλληλεία σε διαφορετική. Ε, πιστεύουμε ότι τροπολογία πιστεύουμε ότι είναι συμβατό να υπάρχει οθολογική διαχείριση της μικρής αυτής αλληλείας και ο καθορισμός των τάκ να γίνεται ανάλογα με το είδος αλληλείας. ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές, βιολογικές πτυχές, αλλά οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πέρας λοιπόν της κοινή συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 11.30. Οπότε συνεχίζουμε με την επόμενη κοινή έκθεση.